Äh, λοιπόν, καλώς ήρθατε. Να περάσουμε στην ημερησία διάταξη με την οποία συμφωνούμε όλοι. Έτσι δεν είναι. Yeah. Wir e di storia This time it's American Express. Check president, you remember? After signing. Soon our voting card will value more. Yeah. Just in case. Wie, gibt es Bemerkungen? Δεν ξέρω αν έχετε... sorry. έχετε παρατηρήσεις. Λοιπόν, καταρχάς να ευχαριστήσω τους Κιώδης και τους συνεργάτες τους για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε τις τελευταίες εβδομάδες. Ευχαριστώ για την καλή διάθεση για να επιτευχθούν συμβιβασμοί. Ήταν δεδομένοι. Οπότε να περάσουμε στις ψηφοφορίες. Πρώτη, η συμβαστική 5, όπως είναι και λογικό. Υπέρ παρακαλώ. Κατά.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 124 linguistisch, 126, 123 Scheck. Hm? Με ακούτε τώρα, με ακούτε τώρα. Συγγνώμη, έχει κλείσει το μικρόφωνο. Πέραση τη ψηφοφορίες. 27-20 εγκρίνεται. ...126 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 127 υπέρ. Dagegen, Enthaltung abgelehnt. 128 dafür, dagegen, Enthaltung abgelehnt. 129 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 130. Απορρίπτεται. 131 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. Απορρίπτεται. 132 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 133 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 134 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 135 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Dagegen Enthaltung angenommen. Antrag 145 dafür ε, δυστυχώς στην 145, λυπάμαι πολύ. Η 14 συμβαστική υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 15 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 16 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 17 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 216. Η 216 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 217 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 18-19 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 220 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 221 υπέρ κατά εγκρίνεται. Η συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 236 υπέρ κατά απορρίπτεται. Η 19 συμβαστική υπέρ κατά εγκρίνεται. Η συμβαστική 20 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ κατά εγκρίνεται, η 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η συμβαστική 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 238 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, Η 238 ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Τσίμα τσίμα. 50... Λέει χαριτολογώντας ο πρόεδρος. 52 με 9 ήταν το αποτέλεσμα. Πάμε στη 2.39. Όχι, εντάξει, την κάνουμε την 39. 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 41, 2.41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 2.42 μαζί με τη 41 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Το άλλο καταπίπτει. Η 244 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 245 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 246 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. η 247 καταπίπτει, η συμβαστική 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η συμβαστική 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, Η συμβαστική 28 υπέρ κατά εγκρίνεται. Η συμβαστική 29 υπέρ κατά εγκρίνεται. Η συμβαστική 30 υπέρ κατά εγκρίνεται. Η συμβαστική 31 υπέρ κατά εγκρίνεται. Η συμβαστική 32 υπέρ κατά εγκρίνεται. Η συμβαστική 33 υπέρ κατά εγκρίνεται, συμβαστική 34 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 35 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 36 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, Συμ... μισό λεπτό, η συμβαστική 37 υπέρ, δύο λεπτά για την τριάντα, η κυρία Γκόμες. Πρόεδρε, υπάρχει αναφορά στον αγώνα ε, κατά των αυξημένων τρομοκρατικών δραστηριοτήτων. Υπάρχει όμως και μία αναφορά ε, στους καταβλισμούς ε, που έχουν σχέση με την τρομοκρατική τρομοκρατικές επιθέσεις. Εδώ υπάρχει μια ανισορροπία. Ή θα πούμε στη, στα κατεχόμενα της Δυτικής Σαχάρας ή θα τα αφήσουμε γιατί τα υπόλοιπα υπάρχουν. Γιατί δεν ξέρω αυτό. Να προτείνω το εξής. Είτε θα ε, διαγράψουμε την αναφορά στους καταβλισμούς ή θα πείσουμε στα κατεχόμενα, στους κατεχόμενους, ε, στα κατεχόμενα εδάφη της Δικής Σαχάρας. Πρόεδρος, εγώ νομίζω ότι υπάρχουν και άλλοι καταβλισμοί και επειδή δεν μπορούμε να τους απαριθμίσουμε όλους, εγώ λέω να διαγράψουμε την αναφορά στους ε, καταβλισμούς. Εντάξει, συμφωνείτε. Λοιπόν, εγώ λέω να ε, δεχτούμε αυτή την... Ε, να ψηφίσουμε χωρίς αναφορά στους καταπλησμούς in doof, όπως λέμε. Λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε τώρα στη συμβαστική 38. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 39. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 41 τη συμβιβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, τροπολογία 4.30 μισό λεπτό υπέρ εγκρίνεται, 450 υπέρ εγκρίνεται, 451 υπέρ κατά εγκρίνεται, Συμβαστική 42. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται η τροπολογία 461. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται η συμβαστική 43. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Κύριε φωνόρντε, μήπως έχετε αφήσει ανοιχτό το μικρόφωνο σας, γιατί σας ακούω συνέχεια στα αυτιά μας. Τα αγγλικά σας είναι πάρα πολύ καλά. Πάμε στην 45, 2.45, υπέρ κατά γκρίνεται. 4.76 υπέρ κατά αποχές 4.81 υπέρ κατά απορρίπτεται. Η 4.82 υπέρ κατά απορρίπτεται. Η 4.83 υπέρ κατά αποχές Το επόμενο καταπίπτει. Πάμε στην 490. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τα επόμενα καταπίπτουν όλα. 494 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 495 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Όχι, μισό λεπτό. Εδώ ηλεκτρονική επαλήθευση για την 495. Έκλεισε η ψηφοφορία. 28 με 25 εγκρίνεται. 496 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 497 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 498 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 500 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 501 ε, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 502 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 503 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 504 υπέρ, κατά, ξανά. Γιατί 504 υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές απορρίπτεται. Η 505 υπέρ, Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται 26 υπέρ 27 κατά. 506 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η άλλη καταπίπτει. 508 υπέρ. 508 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Βλέπω λοιπόν απορρίπτεται 25 υπέρ, 29 κατά. Συμβαστική 46 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 47 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Οπότε περνάμε στη συμβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 44 μετά. Πώς είπατε? Τι είπατε? Who is against block vote? Ποιος είναι κατά του να ψηφιστούν όλες μαζί. Α, οι σοσιαλιστές. Ποιοι είναι κατά της, να ψηφιστούν μαζί μέχρι και την 52. Μα ψηφίσατε, δεν ζητήσατε. Εγώ δεν ζήτησα να ψηφίσετε. Α, καλά, α, καλά. Έγινε δεκτό. Από τις 44 μέχρι την 52. Α, δεν το δέχεστε. 44 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ κατά αποχές έλεγχος.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 Ε, εντάξει, θα μπορούσαμε να το έχουμε ψηφίσει όλα μαζί. Λοιπόν, συμβαστική 3 υπέρ. Κατά απόχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά απόχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά απόχέ, εγκρίνεται. 2 και 3 υπέρ. Κατά απόχέ, απορρίπτεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6, 7, 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 10 α είναι γλωσσική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά αποχές ε, νομίζω ότι εγκρίθηκε. 16 υπέρ. Α, έλεγχος, έλεγχος, εγκάλα. Ελέγχουμε τη 15. Πέρας. 29 υπέρ, 25 κατά και μία αποχή εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 20 εντάξει. Μπούτζα. Όλοι οι συμβιβασμοί καταπίπτουν λόγω της 46 και λόγω της ε, συμβαστικής 47 της Κούλτ. Λοιπόν, τελική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται η έκθεση. 41 ψήφοι υπέρ, 9 κατά, 4 αποχές. 41 ψήφοι πέρα. Ο εισηγητής ε, συγχαίρει τον εαυτό του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Hm? But we have to introduce it. Hmm? Yeah? For Lösing. Hmm? E Η GUE έχει ε, υποβάλει μια έκθεση μειοψηφής και την έχει ήδη στείλει στο γραμματέα. Στη γραμματεία ίσως. Σας ευχαριστώ πολύ. Την έχουμε ήδη λάβει. Την έχουμε ήδη λάβει. Η επόμενη συνεδρίαση μπορεί να είναι την ερχόμενη Δευτέρα. Τρίτη, Α, καλά, τρίτη.